Άλλουσα την προφορική αυτή Κυρία Περφός Πεχές, πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματο τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό μα Κοινοβούλιο υπό την εισηγεσία του κυρίου Γκοζέ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα ενιαίων πληρωμών σε ευρώ. Όταν γινόταν η πρώτη συζήτηση για το σύστημα αυτό, θέταμε ορισμένα ερωτήματα. Σήμερα καταλαβαίνουμε τα ερωτήματα αυτά ήταν θεμητά. Λέγαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ανησυχίες διότι δεν είχαμε την εντύπωση ότι ο ρυθμός κινητοποίησης που ήταν δυσανάλογα μικρός σε σχέση με την κρίση ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Αν θέλουμε το σχέδιο αυτό που, για το οποίο ενδιαφέρθηκαν πολλοί οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα και οι νομοθέτες αλλά που επίσης και κυρίως πρέπει να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο πληρωμών και προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα του ενιαίου νομίσματός μας που αν δεν με λέγεται ευρώ ε, πρέπει να υπάρξει μία κρίσιμη μάζα για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα έχει αποτελέσματα. Ανησυχούμε λοιπόν ιδιαίτερα γιατί οι αυτόματες πληρωμές του σχεδίου ΣΕΠΑ που είναι από τις πιο πρωτοπόρες πτυχές του συναντούν ακόμη δυσκολίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι ως προς την ευθύνη της Κομισιόν τίθενται δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς σκοπεύει να προωθήσει και να στηρίξει τη μεταβολή των συνήθων διαδικασιών πληρωμών στο καινούριο ΣΕΠΑ. Τα λαμβάνει υπόψη της όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας, αν αμφιβάλλουμε και συμφωνεί ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα μια κρίσιμη μάζα που να έχει μεταφερθεί στο ΣΕΠΑ μέχρι το 2010. Αλέως τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί αυτό. Δεν προβλέψαμε καμία δεσμευτική ημερομηνία για την υποχρεωτική μεταφορά των μηχανισμών πληρωμών στο ΣΕΠΑ. Καιρό θα ήταν όμως να γίνει κάτι τέτοιο ο καθορισμός αυτός. Γιατί υπάρχουν ακόμη κενά ως προς τη συμβατότητα των υπαρχόντων συστημάτων με το μελλοντικό ΣΕΠΑ. Πράγμα που εμποδίζει τη μεταφορά τους. Και γι' αυτό νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να βοηθήσει τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα θεμητά αυτά ερωτήματα. Έπειτα υπάρχει και το θέμα των προμηθειών που έχει παραγνωριστεί ενώ για πολλούς επιχειρηματίες είναι ένας από τους όρους για την επιτυχία του σχεδίου ΣΕΠΑ. Καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι οι διάφοροι ηθήνοντες, δηλαδή είτε από τον τραπεζικό τομέα είτε από τη διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Καιρό θα ήταν να αναλάβουν όμως όλοι τις ευθύνες τους. Γιατί θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ένα μηχανισμό που έχει κάποια συνέπεια χωρίς να δώσουμε τους παράγοντες της αγοράς αυτής και τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει δηλώσει ότι υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού, ότι αντιτίθεται η διάταξη αυτή στους κανόνες του ανταγωνισμού, αλλά δεν μας έδωσε καμία εναλλακτική λύση, ενώ ούτε έχει δοκιμαστεί καμία. Άρα δεν ξέρουμε αν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι σε θέση να προβλέψει εναλλακτικές λύσεις που να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά μας. Παράδειγμα, η χρηματοδότηση ενός euh, du τέτοιου συστήματος που να βασίζεται στην ταύτιση των παραβιάσεων που θα έχουν σημειωθεί δεν μου φαίνεται κάτι το λογικό ούτε το δίκαιο κοινωνικά. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή δύο πράγματα ζητώ. Να ορίσει μια τελική ημερομηνία για τη μεταφορά και να βοηθήσει να καθοριστεί ένα εναλλακτικό σύστημα ή τουλάχιστον αποδεκτό γενικά με όρους συνθήκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Μπερβάνης Σπυρές. και τώρα η κυρία Επίτροπος Ανδρούλα Βασιλείου. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξέρουμε Καταρχήν θα ήθελα να σας μεταβιβάσω το, ε, ε έτσι συγγνώμη του Επιτρόπου Μακρύβη που δεν μπορούσε να είναι παρόν. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εξετάζεται, γιατί και η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα για τον εφαρμογή του ΣΕΦΑ σοχνά, σοχ, σωστά αναφέρει τα κύρια θέματα που πρέπει να εξεταστούν για τη σωστή εφαρμογή του ΣΕΠΑ. Πρώτον, πώς σκοπεύει η Κομισιόν να προωθήσει την μετάφαση μέσα του ΣΕΠΑ. Το ΣΕΠΑ είναι ένα προϊόν που προωθείται από την αγορά. Αλλά λόγω του ωφέλου του για την ευρύτερη οικονομία, η Κομισιόν προσπάθησε να προωθήσει τη μετάβαση, παραδείγματο χάρη δρώντας ως καταλήτης για να αυξηθεί το πολιτικό προφίλ του ΣΕΠΑ μέσω μιας έκθεσης για το ε, ΣΕΠΑ και προωθώντας την μετάβαση των δημοσίων ορχών. Okay. Επίσης ε, προσπαθώντας ίδια να υιοθετήσει έγκαιρα το ΣΕΠΑ και τέλος όπως ελέγχθη την τελευταία εβδομάδα στην δημοσία της Κομισιόν για την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης Ευρώπης ότι πρέπει να φροντίσουμε να πραγματοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του ΣΕΠΑ. Κατόπιν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα έχει πραγματοποιηθεί πλήρωση η μετάβαση αυτή μέχρι το 2010. Προσπαθούμε να περιορίσουμε το κόστος βέβαια, παρόλο που ε, επιτυχώς ε, ξεκίνησε ε, το ΣΕΠΑ, λιγότερο από το 2% των πληρωμών έχουν μεταφερθεί. Ε, επίσης, ε, ο σημερινός ρυθμός της μετάβασης είναι πολύ μικρός για να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα μέχρι το 2010. Το τρίτο θέμα ήταν για την αναγκαιότητα σαφής και δεσμευτικής καταληκτικής ημερομηνίας. Ναι, ναι. Βλέπουμε πόσο χρειάζεται να οριστεί μια τέτοια ημερομηνία. Βέβαια, 2012 δεν φαίνεται και παράλογο. Παρ' όλα αυτά, για πολλά κράτη-μέλη αυτό εξακολουθεί να είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ του ορισμού μίας διαδικασίας για να εξεταστεί το θέμα συλλέγοντες πληροφορίες για τις επιπτώσεις μιας καταρρεκτικής ημερομηνίας στους διάφορους ενδιαφερόμενους και έχοντας μία εις βάθος συζήτηση μαζί τους. Αυτό ίσως ε, προετοιμάσει την οδό για πολιτική υποστήριξη και αν χρειαστεί ενδεχόμενη νομοθετική πρόταση παραδείγματος χάρη στα τέλη του έτους. Το τέταρτο ερώτημα λέει πώς θα υπάρχει νομική ασφάλεια για το ΣΕΠΑ σε σχέση με το MIF. Εμείς χρειάζομαστε να υπάρχουν νομική ε, σαφήνεια για να μπορέσει να προωθηθεί επιτυχώς η οδηγία για το ΣΕΠΑ. Και γι' αυτό η Κομισιόν υποστηρίζει πληρώσει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ναι. για να εξευρηθεί μια προσωρινή απάντηση μέσα στα πλαίσια της αναθερώτησης του κανονισμού για τις ε, διασυνοριακές πληρωμές. Η Κομισιόν υποστηρίζει επίσης ε, να υποστηριχτεί η νομική η ισχύ της, των εθνικών διατάξεων για τη μετάβαση στο ΣΕΠΑ. Αυτό βέβαια είναι νομικό θέμα που θα πρέπει να επιληθεί από τις εθνικές αρχές. Παραδείγματο χάρη χρησιμοποιώντα τη δυνατότητα που δίνουν οι οδηγίες για την πληρωμή των υπηρεσιών. Το πέμπτο ερώτημα αφορά το πώς η Κομισιόν εξετάζει το θέμα του MIF για πληρωμές με κάρτες. Αυτό το θέμα προωθείται κυρίως μέσω της αξιολόγησης της Κομισιόν των δύο κυρίων διεθνών ε, καρτών, Mastercard δηλαδή και Visa. Το Δεκέμβριο του 2007 η Κομισιόν αποφάσισε ότι το Mastercard MFS δεν ήταν συμβατό με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Η Mastercard έχει προσφύγει κατά της απόφασης Κομισιόν. Το Μάρτιο του 2008 η Κομισιόν εκείνη το τη διαδικασία για να δει κατά πόσον η Visa και το MIF της Ευρωπαϊκής είναι ε, μια παράβαση του άρθρου 81. Οι ζητήσεις με τη Visa συνεχίζονται επίσης η Κομισιόν προσπαθεί να ε, επιτύχει ένα ισοπεδίο ο παιδής για την κάθε τη Visa και οποιασδήποτε άλλες κάρτες προσωστούν στο μέλλον. Η πρώτη αυτή σα ερώτηση ε, ρωτάει κατά πόσο η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει μια τελική πρόταση για το θέμα MIF σε μια οικονομία αγοράς η βιομηχανία είναι εκείνη που θα πρέπει να υποβάλει ε, το κατάλογο μοντέλο. Όπως σας είπα για τις ε, πληστορικές συνεχίζεται να συζητήσει αυτή τη στιγμή με την Mastercard και με τη Visa. Όσον αφορά για το άμεσο ε, κόστος η, Κομισιόν θέλει μέσω του εν λόγω, κλάδου να βοηθήσει δίνοντας ως πλήρη στοιχεία και φροντίζοντας να συμβάλλουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στην αγορά. Αυτό θα πρέπει να πετυχθεί το αργότερο τον Νοέμβριο του 2009. Τελευταίο σας ερώτημα. Τελευταίο ρωτάτε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που σκοπεύει η Κομισιόν να προτείνει ούτω ώστε η μετάβαση στο ΣΕΚΒΑ να είναι οδηγήσει σε πιο ακριβά συστήματα πληρωμών. Σήμερα την από τη Κομισιόν αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Πρώτον, η ΣΕΒΑ θα πρέπει να προωθήσει τον οργανισμό και να αυξήσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω οικονομιών ε, μεγάλων διαστάσεων που και τα δύο θα οδηγήσουν σε πίεση του κόστους προς τα κάτω. Επίσης θα πρέπει να προστατευτούμε από την επικάλυψη του κόστου, από το κρυμμένο κόστος, παρόλο που ίσως ορισμένοι κατανοτές θα δίνουν ότι η τιμή αυξάνεται μεν, αλλά εκείνοι μεταβαίνουν από υψηλό ε, από καλυμμένο κόστος σε πραγματικό κόστος εις τους. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μια σειρά μελετών και τέλος συμφωνήσαμε ότι υπάρχει μια ανησυχία από τελεσματικά εθνικά προγράμματα πιστοτικών καρτών μπορούν να αντικαταστούν ίσως από άλλα εναλλακτικά ε, συστήματα θα μπορούσαμε ίσως να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα καρτών debit και έτσι, εν καταλήξει, η ΣΕΠΑ θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών και ε, επαρκώς ασφαλής κάρτες με στα πλαίσια της ε, κοινοτικής πολιτικής. Όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό χαιρετίζω την ε, το ε, ψήφισμα αυτού και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για το ΣΕΠΑ. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε κυρία μου. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Για τρία λεπτά, Γκοζές ε, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά ακούσαμε για την οδηγία αυτή για τις πληρωμές ε, για την οποία ήμουν εισηγητή στο Κοινοβούλιο και επενεκτήθηκα την πρώτη ανάγνωση του 2007. Η οδηγία αυτή οδήγησε τον τραπεζικό τομέα να διαθέσει τα κατάλληλα, να διαθέσει τα κατάλληλα νομικά εργαλεία για να εφαρμοστεί το σχέδιο ΣΕΠΑ για τις πιστοτικές κράτες, ε, κάρτες και τις υπόλοιπες πληρωμές σε ευρώ τελικά δεν θα υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ εθνικών και διεθνών πληρωμών. Και αυτό θα έχει πλεονεκτήματα και για τον τραπεζικό τομέα και για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Προσέξαμε τα εργαλεία του σχεδίου ΣΕΠΑ να μην έχουν σαν επίπτωση περισσότερο κόστος για τον πολίτη. Από την έγκριση της έκθεσής μας μέχρι τώρα τα πράγματα προχώρησαν υπερβολικά αργά. Τον Οκτώβριο του 2008 μόνο 1,7% των πληρωμών γινόταν, γίνονταν σύμφωνα με το σχέδιο ΣΕΠΑ. Και γι' αυτό σήμερα εγκρίνουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει από την Κομισιό να καθορίσει μια υποχρεωτική ημερομηνία μέχρι την οποία να έχουν μεταφερθεί όλες οι πληρωμές στο σύστημα αυτό. Όχι όμως μετά το Δεκέμβριο του 2012. Πριν γίνει η μεταφορά αυτή βέβαια, πρέπει να διακανονιστεί το λεπτό πρόβλημα των προμηθειών. Δεν πρέπει να καταργηθούν. Οι υπηρεσίες πληρωμών είναι και αυτές μία εμπορική δραστηριότητα που εμπεριέχει κάποιο κόστος και κάποιο θεμητό κέρδος. Αντίθετα πρέπει να αποφύγουμε την έλλειψη διαφάνειας ή την αυθαιρεσία. Πρέπει να καθοριστούν λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές για τις προμήθειες αυτές. Και για περισσότερη νομική ασφάλεια πρέπει οι αυτέ αυτές γραμμές να αναγνωριστούν από όλου πριν αρχίσει η πλήρη εφαρμογή του ΣΕΠΑ για τι πληρωμές. Χωρί αυτή τη νομική διασφάλιση οι τράπεζε πολλών χωρών δεν θα εφαρμόσουν το νέο σύστημα των πληρωμών και μπορεί και να υπάρξει και παράλυση του. Το ΕΛΚ και το ΕΣΚ εξάλλου κατέθεσαν τροπολογίες πολύ παρόμοιες μεταξύ τους για την αυριανή ψηφοφορία και προφανώς ε, θα θέλαμε να εγκριθούν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κουσιαστή. Τώρα θα αρχίσει η διαδικασία της οφθαλμοθυρίας. Η κυρία Στάκεβιτ πρώτα. Για δύο λεπτά. Έχετε το λόγο κύριε. μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας στα χέρια μας. Αυτό θα ήταν και μια πηγή νέων μέτρων. Σήμερα συζητάμε το θέμα της αγοράς πληρωμών. Είναι πραγματικά λυπηρό που οι λύσεις μας πραγματοποιούνται τόσο διστακτικά ένας λοσυγματικός λόγου λέγεται ότι δεν έχουν οι τράπεζες επαρκείς ε, τεχνικές δυνατότητες. Αλλά ομολογώ ότι ο τεχνικός εξυγχρονισμός των τραπεζών είναι προς όφελος και της ίδιας της τράπεζας. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουν τις αγορές τους, τις μεθόδους πληρωμής τους, για να μπορέσουν να κερδίζουν και περισσότερα από όλα αυτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι συμμετέχουν σε αυτούς τους κλάδους να είναι πιο αποτελεσματικοί και να είναι πιο αποφασισμένοι στη μετάβαση προς το ΣΕΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ο κύριος Ρούμπικ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι. Ξέρουμε ότι ο νέο Ευρωπαϊκό Χώρο πληρωμών είναι μια πραγματική πρόκληση ιδίω για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις γιατί αυτοί εργάζονται πολύ έντονα με τα συστήματα επιστοτικών κρατών και το κόστος της χρήσης του συστήματος αυτού είναι πολύ διαφορετικό. Θεωρώ εδώ λοιπόν ότι η ε, διαφάνεια δεν προσφέρεται επαρκώς. Ιδίω μέσα στα πλαίσια μας κρίσης χρειαζόμαστε για τις επιχειρήσεις μια επαρκή ενίσχυση. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να αυξηθεί η αξιοπιστία των επιχειρήσεων και θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει αυτό με το ΣΕΠΑ για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ωφεληθούν μόνο οι μικρές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ότι οι σχέσεις μικρών και μεγάλων θα είναι πιο αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπικ. Το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Φασιλείου. I θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και την ε, Πρόεδρό της, την κυρία Περβάνς Περές, για την συζήτηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΣΕΠΑ, ε, το οποίο δεν είναι μόνο μια πρωτοβουλία αυτορύθμισης, αλλά πρόκειται και για μια ε, βασική ρύθμιση η οποία ενισχύει την νομισματική ένωση, όπως επίσης και τη στρατηγική της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σαφώς έχουν το ίδιο όραμα και το ίδιο στόχο για το ΣΕΠΑ. Να σας ε, υπενθυμίσω όμως τρία βασικά σημεία. Πρώτον, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην προσπάθειά της να γίνει η μεταφορά της διαδικασίας ε, του ΣΕΠΑ ε, μέσω πίεσης προς τις δημόσιες αρχές για ε, να την εγκρίνουν το νωρίτερο δυνατόν. Και θα συνεχίσουμε ανελαίητα τις προσπάθειές μας ε, για την εφαρμογή του ΣΕΠΑ. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι ότι συμμεριζόμαστε την, ε, ε, το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ενημέρωση του ΣΕΠΑ, δεν θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αυτή τη στιγμή και είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται πολύ βασική εργασία πριν αναλάβουμε ε, μια τέτοια δέσμευση. Τρίτον, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει ε, κατευθυντήριες γραμμές για την ε, βασική ε, αποζημίωση και τον συμβιβασμό τους με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ξέρουμε ότι υπάρχει λίγος χρόνος μέχρι την θέση σε εφαρμογή της άμεσης χρέωσης του ΣΕΠΑ και θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα τα κατευθυντήρια στοιχεία πριν από τον Νοέμβριο του 2009. Να εμείνω όμως σε ένα στοιχείο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να δοθούν εάν και μόνο αν ο κλάδος μας δώσει συγκεκριμένες ιδέες για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα επιχειρησιακά μοντέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Βασιλείου. Λάβαμε μια πρόταση ψηφίσματος ε, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ε, η οποία θα ψηφιστεί αύριο στις 12 να ε, περάσουμε τώρα μετά από τη λήξη αυτής της συζήτησης στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη το οποίο προβλέπει τη συζήτηση για ένα μια πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα. Περιμένουμε την ε, κυρία Επίτροπο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο